11 περίπου. Επόμενο θέμα. Επόμενο θέμα. Εδώ. Είναι προφορική ερώτηση για την μεσοπρόθεσμη χρηματοοικονομική βοήθεια για τα εισαζύγια πληρωμών των κρατών μελών και τις κοινωνικές προϋποθέσεις. Από τρεις βουλευτές τριών πολιτικών ομάδων. Πρώτα, για δύο λεπτά, η κυρία Τατιάνα Ζντανόκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι. Προέρχομαι από την Λετωνία, μια χώρα που επλήγει σοβαρά και θα είχε χρεοκοπήσει χωρίς βοήθεια από το εξωτερικό. Ε, πήραμε βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνέ Νομισματικό Ταμείο έπρεπε όμως να περικόψουμε τον προπολογισμό μας ως προϋπόθεση και αυτό το έκανε μειώνοντας τις συντάξει κατά 10% και 70% των συνταξιούχων που εργάζονται και μείωσε τα οικογενειακά επιδόματα κατά 10% και μείωσε επίσης και το φορολόγητο όριο. Όπως βλέπετε ήταν ε, τελείως ίδια η προσέγγιση, είτε η σύνταξη ήταν 100 ευρώ είτε 1000, 10% περικοπή. Η Κομισιόν καλωσόρισε αυτές τις σκανδαλώδεις ε, περικοπές ε, στο μνημόνιο με την Λετωνία. Ήταν σαφές ευθύς εξ αρχής πως τέτοιες γενικές περικοπές θα έπληκαν τους πιο ευάλωτους. Την ε, παραμονή τέτοιων σημαντικών ε, γεγονότων. Και η Ουγγαρία και η Ρουμανία έλαβαν ανάλογη βοήθεια. Δημιουργείται έτσι ένα προηγούμενο για την αποδοχή άδικων κοινωνικών μέτρων που δεν πρέπει να γίνει. Βεβαίω, κύριε Επίτροπε, θα πείτε πω εμεί τα λεφτά δίνουμε και η κυβέρνηση μετά εφαρμόζει την κοινωνική πολιτική. Όμω, τα κοινωνικά δικαιώματα είναι δεσμευτικά για τα θεσμικά όργανα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη του τα θεσμικά όργανα. Αλλιώ τα λόγια που λέμε για υψηλό επίπεδο κοινωνική ε, προστασία θα κάνουν του ανθρώπου να υπομοιδιούν ηρωνικά. Ευχαριστούμε. Για δύο λεπτά η κυρία Λίν έχει τον λόγο. Εδώ δεν πρόκειται να καθορίσουμε εμείς τι θα κάνει κάθε χώρα και πώς θα δαπανίσει τα χρήματά της. Η κάθε χώρα έχει δικές της μεθόδους για να βγει από την οικονομική κρίση. Όταν όμως χορηγείται βοήθεια της Ένωσης για τον σκοπό αυτόν θα πρέπει να δαπανούν τα κονδύλια με τρόπο που να σέβεται τις αρχές της Ένωσης. Να μην αγνοεί δηλαδή την ανάγκη και για κοινωνική προστασία. Η οικονομική αυτή κρίση έπληξε τους πολίτες ολόκληρης της Ένωσης και γι' αυτό είναι σωστό που υπάρχει αυτό το ταμείο. Πολλοί έχασαν τη δουλειά τους και κατέληξαν ως άνεργοι να είναι από τους πιο ευάλωτους πολίτες. Δεν πρέπει να τους αγνοήσουμε και αυτό πρέπει να φαίνεται. Ιδιαίτερα πρέπει να μας ενδιαφέρει, με ενδιαφέρει να μάθω, εάν οι χώρες είναι υποχρεωμένες να αναφέρουν στην Κομισιόν και κατά πόσον σεβάστηκαν αυτή την κοινωνική διάσταση στα προγράμματά τους. Είναι σημαντικό να δώσουμε το σωστό μήνυμα στις χώρες που παίρνουν ενωσιακά κονδύλια. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να αποσαφινιστεί ότι η Κομισιόν θα μπορούσε να λάβει υπόψη της και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να βοηθηθούν περισσότερο και καλύτερα οι ασθενέστεροι πολίτες. Ξέρω ότι υπάρχουν οικονομικές δυσκολίες αλλά και ότι μάλλον δεν είναι εύκολο να λάβει κανείς πάντοτε υπόψη του τις κοινωνικές συνέπειες των μέτρων αλλά δεν πρέπει και να το ξεχνάμε διότι η οικονομική κρίση έχει και ανθρώπινο πρόσωπο και το πρόσωπο αυτό εκπροσωπείται συνήθως από τους επαναλαμβάνω ασθενέστερους πολίτες. Ευχαριστούμε κύριε Αλήν. Για δύο λεπτά ο κύριος Θέρκας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Πριν υποβάλω το ερώτημα Διάβασα πολύ προσεκτικά τα προηγούμενα και παλαιότερες θέσεις που είχε λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από αυτού του θέματος. Και είναι γεγονός ότι στις 23 Απριλίου του 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκρινε μια νομοθετική πράξη για τροποποίηση του κανονισμού 2002 που σύμφωνα με το άρθρο 100 ε, ρυθμίζει την διψηνοϊκή κατάσταση. Και αυτό το ψήφισμα κύριε Πρόεδρε ε, ξέφρασε τη θετική του άποψη το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ρυθμιστούν τα συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κράτη που πλήττονται από την κρίση εκφράζει σαφώς την αλληλεγγύη του για τα πλέον πρόσφατα προσχωρήσαν τα κράτη στην Ένωση. Λέει όμως επίσης ότι αυτές οι ενισχύσεις θα πρέπει να πληρούν τέσσερα κριτήρια. Ποιοτική δημόσια δαπάνη, όχι διασπάθηση δηλαδή των πόρων, Δεύτερον, αηφορία. Τρίτον, πολιτική πλήρους απασχόλησης. Και τέταρτον, καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Είναι προφανώς στόχοι που θα πρέπει να γίνουν απανταχού σεβαστοί. Από ΜΚΟ, από συνδικάτα, από πολίτες έγιναν δεκτά όλα αυτά. Και αυτά τα κράτη, υπάρχουν κράτη τέλο πάντων που έχουν λάβει πολύ σημαντικά και ψηλά ποσά. Και όπω έλεγε η συνάδελφο, έχουν περικοπεί 40% στην εκπαίδευση, 30% για τα εισαδεξιοδότηση, 50% οι επιχορηγήσει για του ασθενεί. Έναντι αυτή τη πραγματικότητα, ε, κύριε Πρόεδρε, το Κοινοβούλιο επιθυμεί τουλάχιστον η σιωπή μα να μην ερμηνευθεί ω ε, συνένεση ότι επιβάλλουμε και εμεί αυτά τα μέτρα, ότι συνενούμε. Όχι, δεν είμαι θα συνενοχή στην διάπραξη αυτού του αδικήματος. Δεν είναι δυνατόν ποτέ να δεχθούμε την ε, νύφη να την πληρώσουν οι πιο αδύναμοι. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος Αλμούνια. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες ε, και κύριοι Ευρωβουλευτέ. Τα προβλήματα στην Λετωνία, την Ουγγαρία και την Ρουμανία που είναι οι τρεις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που λαμβάνουν ε, δάνεια μέσω της διευκόλυνσης ισοζύγιο πληρωμών δεν τα δημιούργησε ούτε αυτό το Κοινοβούλιο, ούτε η Κομισιόν, ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονομική κρίση τα δημιούργησε. Απλώς τα αποτελέσματα έγιναν οξύτερα, τα προβλήματα έγιναν οξύτερα από κακοδιαχείριση των υπευθύνων αυτών των χωρών. υπάρχουν και άλλες χώρες στην ίδια ευρύτερη περιοχή με αυτές που δεν έχουν τα ίδια προβλήματα και που μπορούν να αντιμετωπίσουν την κρίση με πολύ καλύτερες συνθήκες. Με ενίσχυση βεβαίως από τα ευρωπαϊκά κονδύλια, ταμείο συνοχής, διαθωτικά ταμεία, με την προπτική να ενταχθούν στο ευρώ, αλλά χωρίς να απολάβουν αυτής εδώ της ενίσχυσης, της συγκεκριμένης. Γιατί Λοιπόν, και γιατί αναγκαστήκαμε για τις άλλες χώρες να δανείσουμε χρήματα. Όχι επειδή φταίμε εμείς, αλλά επειδή εκείνοι, οι υπεύθυνοι αυτών των χωρών, τα θαλάσσωσαν εις ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος. Δανείζουμε, αλλά κανένας δανειστής δεν δανείζει χωρίς προϋποθέσεις. Βάζουμε λοιπόν προϋποθέσεις και μάλιστα σκληρές και αυστηρές και λέμε σε αυτές τις χώρες δεν θα λείψουν χρήματα για να συγχρηματοδοτήσετε διαρθρωτικά ε, μέτρα αλλά μην περικόψετε δινερό μην ε, περικόψετε συγγνώμη χρήμα από τους πιο αδύναμους μην περικόψετε χρήμα για τις μεταρρυθμίσεις εγώ συμφωνώ με τις δικές σας ανησυχίες και όχι μόνο τις συμμερίζομαι αλλά εγώ, όπως και εσείς φαντάζομαι, τις διαβιβάζω και στους πολιτικούς ηθήνοντες. Τρία δις. Τρία δις. Για τη Λετωνία. Πολύ σημαντικά ποσά για την ε, Ουγγαρία. Και προσοχή. Κανείς δεν δανείζει χωρίς προϋποθέσεις. Το ξανάπα. Δεν μπορούμε να λάβουμε αποφάσεις όμως που είναι ευθύνη των κοινοβουλίων και των κυβερνήσεων αυτών των χωρών. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να επενθυμίσουμε τις παραμέτρους ε, στους ηθήνοντες. Την ευθύνη που έχουν να βγάλουν τους πολίτες τους από την κρίση. Και δύο, τους υπενθυμίζουμε ότι για μέτρα που υπερβαίνουν το απολύτως απαραίτητο δεν θα λάβουν κονδύλια. Διότι θα πρέπει να σταθούν τα, στα πόδια τους χωρίς δεκανίκια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε και τώρα θα μιλήσουν οι εκπρόσωποι των ομάδων μέρους του ΕΛΚ, ο κύριος Γοζές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτά που είπε ο Επίτροπος είναι μια πραγματική απάντηση στο ερώτημα που τίθεται εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χορηγεί κονδύλια χωρίς όρους και οι όροι τους όρους υπενθύμησε ο Επίτροπος βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτική απασχόληση, αντιμετώπιση κλιματολογικών ελλαγών αλλά και η αναγκαιότητα ανταπόκρισης ως το δυνατόν συντομότερα στις ανεπάρκειες της εσωτερικής διαχείρισης ώστε οι χώρες τις οποίες βοηθούμε να μπορούν να φτάσουν σε, στο αρμόζον επίπεδο. Δεν πρέπει όμως να υπερβάλλουμε στην, όταν θέτουμε όρους. Πρέπει να δείξουμε κάποια εμπιστοσύνη και στις χώρες που λαμβάνουν την οικονομική βοήθεια της Ευρώπης για να μπορέσουν να πάρουν τα μέτρα που χρειάζονται και να μην ληφθούν, να μην ληφθούν μέτρα που δεν ε, συμφωνούν με την πραγματικότητα όπως είπε και ο Επίτροπος. Πρέπει επαναλαμβάνω στα, και στα κράτη-μέλη να επιδειχθεί η απαραίτητη εμπιστοσύνη ώστε να ορθοποδήσουν και να μην γίνουν εξονυχιστικοί και άχρηστοι έλεγχοι που δεν θα φέρουν κανένα αποτέλεσμα. Οι καινούργιες επιχορηγήσεις που μπορεί να εγκριθούν θα φανεί τι επιπτώσεις είχαν και ποια μέτρα ήταν τα κατάλληλα και ποια δεν ήταν, ιδίως στο κοινωνικό τομέα. Ευχαριστούμε κύριε Γκοζές. Τώρα εκ μέρους των σοσιαλιστών η κυρία Μπέρετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα το θυμόσαστε. 24 Απριλίου το υπενθύμισε ο Αλεξάνδρ Σέρκας όταν ε, δεχτήκαμε, επικυρώσαμε ε, την ε, διευκόλυνση αυτή για το ισοζύγιο πληρωμών, το κάναμε υπό δύο προϋποθέσεις. πρώτη προϋπόθεση είναι οι σχέσει αυτές να συνοδεύονται από προϋποθέσεις κοινωνική κυρίω φύσεω. Και δεύτερον, να υπάρχει διαφάνεια εναντί αυτού του Κοινοβουλίου ει ό,τι αφορά τι συνθήκε επί τι οποίε τέτοιε συμφωνίε συνάπτονται με τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι η σημερινή συζήτηση είναι σωστή, χρήσιμη και δημοκρατική αρκεί βεβαίως να συνοδευτεί και από αποτελεσματικότητα. Λοιπόν, ε, υπάρχει κρίση η οποία θέτει να αμφιβόλω και τις θεμελιώδεις αρχές την ε, αλληλεγγύη έναντι των κρατών μελών έναντι ορισμένων κρατών μελών και τα νέα που έρχονται από τη Ρουμανία μόνο επιβαρύνουν, επιδεινώνουν αυτή την κατάσταση λόγω της πολιτικής ε, αβεβαιότητας που υπάρχει μετά τις συνέπειες αυτής της κρίσης, αλλά και άλλους παράγοντες. Έχουμε τεράστιες δυσκολίες. Δεν θα ήθελα να αναπαραγάγουμε όμως εδώ τα λάθη του παρελθόντος και ιδίως αυτά τα οποία χαρακτηρίσαμε τα λάθη του Δουνουτού, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου δηλαδή, που έκανε το κακό χειρότερο με τα μέτρα που ενέκρινε ο Ζων Πολ Γκοζές ε, όταν μας λέει να μην κάνουμε εξονυχιστικούς ελέγχους και να περιμένουμε το επόμενο αίτημα για να εξετάσουμε και να ελέγξουμε την ποιότητα της χρήσης της βοηθείας, της ενισχύσεως. Όχι, όχι, όχι, όχι. Τη στιγμή που δεχόμαστε να δώσουμε την ενίσχυση θα πρέπει να κάνουμε τον έλεγχο. Δεν μπορούμε να εθιλοτυφλούμε ή να αγνοούμε την πραγματικότητα ή να κλείσουμε τα όματά μας. Είμαστε, δεν μπορούμε να δεχθούμε οι πλέον ευάλωτοι, όπως είπε κάποιος συνάδελφος, να πληρώσουν την ύφη. Και βεβαίως δεν κατηγορούμε την Κομισιόν για, κακοδιαχείριση της, ε, για την κακοδιαχείριση της λετωνικής κυβέρνησης. Κανείς, ουδής ε, κύριε Επίτροπε, στο κοινοβούλιο αυτό ε, τόλμησε ε, και θα τολμήσει ποτέ να πει κάτι τέτοιο. Αλλά δεν μπορούμε από το δημόσιο κορβανά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ε, βγάλουμε λεφτά για βοήθεια της Λετωνίας τα οποία θα είναι εις βάρος του πλέον ευάλωτου Λετωνού πολίτη και όχι υπέρ της ισορροπίας ε, στην οικονομία και την αγορά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Για δύο λεπτά. Για τους φιλελεύθερους. Η κυρία Χάρκιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η διαδικασία κοινωνικής συνοχής Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πολύ σημαντική αν να επιτύχουμε τον στόχο της διαρκούς ανάπτυξης περισσότερες και καλύτερες δουλειές και περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασία και κοινωνική συνοχή. Υπάρχει κοινωνικό αποκλεισμό για πολλού πολίτε, αλλά ειδικά για αυτού που είναι στο περιθώριο τη κοινωνία, για όσου είναι άνεργοι και για αυτούς που βασίζονται στο κοινωνικό δίκτυο ασφαλείας των διαφόρων κρατών μελών. Το ερώτημα που απευθύνει τη Κομισιόν είναι εάν προσπαθεί να ενσωματώσει την πολιτική κοινωνικής συνοχής όταν δίνει μεσοπρόθεσμη ε, ενίσχυση στα κράτη-μέλη για το ισοζύγιο πληρωμών σύμφωνα με τον κανονισμό 332 του 2002. Εγώ δεν είμαι υπέρ των πολλών όρων και της πολλής γραφειοκρατίας όταν δίνουμε βοήθεια. Είτε μιλάμε για κράτη-μέλη, είτε μιλάμε για άτομα και μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όταν όμως αυτό σημαίνει πώς θα εφαρμόσουμε μια βασική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κοινωνική συνοχή, τότε είναι σημαντική η όρη. Δεν μπορούμε εμείς εδώ πέρα να γράφουμε συνεκώς έγγραφα για το πώς θα επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή και ταυτόχρονα να μην διασφαλίζουμε πώς αυτή η διαδικασία ενσωματώνεται στις πρωτοβουλίες μας. Η Κομισιόν έχει δώσει αυτά τα δάνεια με σκληρούς όρους, αλλά δεν ήταν σαφές ποιοι ήταν αυτοί οι όροι και αν συμπεριλαμβάνουν όντως κοινωνικούς όρους ανεξαρτήτως των ε, συνθήκων εκταμίευσης ε, κοινωνικών κονδυλίων δεν μπορούμε να ανοίπτουμε τα σχήρας μας και να ελπίζουμε για το καλύτερο. Εντάξει, καλό το να εμπιστευόμαστε τα κράτη-μέλη, αλλά πρέπει να κερδίσουν την εμπιστοσύνη μας και αν υπάρχουν ανησυχίες πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε. Ευχαριστώ, κυρία Χάρκιν. Τον λόγο για ένα λεπτό έχει για την ε, ο κύριος Λε Χιουαρικ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε. Οι περισσότεροι οικονομολόγοι διαπιστώνουν ότι η κρίση οφείλεται κυρίως στη μεταφορά πλούτου από την εργασία προς το κεφάλαιο. Και γενικώ συμφωνούν ότι στις χώρες όπου διατηρήθηκαν οι δημόσιες υπηρεσίες και τα συστήματα κοινωνικής περίθαλψης υπέφεραν λιγότερο οι πληθυσμοί τους. Εδώ όμως μας ενδιαφέρει η φύση των όρων που θέτετε για να χορηγήσετε κονδύλια για να βοηθηθούν οι πληθυσμοί αυτοί. Δεν μπορεί να είναι όρος η εφαρμογή διαρθρωτικών προγραμμάτων που μειώνουν τις κοινωνικές δαπάνες και τις δαπάνες για την παιδεία καθώς και τις κοινωνικές υπηρεσίες ή τις δημόσιες υπηρεσίες γενικού συμφέροντος. Όλα αυτά δεν πρόκειται παρά να χειροτερέψουν την κρίση, την ανεργία και την ανέχεια. Γι' αυτό πρέπει νομίζουμε να αντιστραφούν τα κριτήρια και οι όροι και να αποφασιστεί ότι τα ευρωπαϊκά ταμεία ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πρέπει να συνδυάσουν τη χορήγηση κονδυλίων με ένα νέο τύπο δανειοδότησης ώστε να υπάρξει μια νέα κατανομή του πλούτου με σεβασμό του κοινωνικού και κτημένου και της κοινωνικής προστασίας για να υπάρχει εγγύηση εργασίας για όλους και όλες. Γιατί αλλιώς δεν θα εκρόκειται να υπάρξει καμία οικονομική αποτελεσματικότητα. Ευχαριστούμε κύριε Λεαρίκ. Τώρα οι υπόλοιποι. Πρώτος για δύο ολόκληρα λεπτά ο κύριος Καρίνης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Επίτροπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε τις ε, χώρες ε, οι οποίες ε, βρέθηκαν σε δύσκολη θέση με την κρίση. Τα σταθερά κοινωνικά συστήματα δεν υπάρχουν χωρίς σταθερή οικονομία οι συνάδελφοι προτείνουν εδώ πέρα να γίνουν πιο αυστηροί οι όροι της οικονομικής βοήθειας. Δεν είναι σωστό αυτό. Πρέπει να σκεφτούμε μάλλον την διεύρυνση αυτών των κριτηρίων. Δεν πρέπει να δίνουμε βοήθεια μόνο για σταθεροποίηση του προϋπολογισμού αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας. Επενδύσεις στην οικονομία είναι απαραίτητες έτσι ώστε να εγγυηθούμε μακροπρόθεσμα τα κοινωνικά συστήματα. Όλοι αυτοί οι στόχοι πρέπει να ακολουθηθούν από τα κράτη που βρίσκονται σε οικονομικές δυσκολίες. Η αντιμετώπιση της κρίσης και η περαιτέρω σταθεροποίηση συνδέονται στενά με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έναντι των χωρών αυτών. Μόνο έτσι θα έχουμε κάρπους σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίση δεν μπορεί οι χώρες αυτές να βασίζονται μόνο σε ε, τέτοιες ε, ενισχύσεις πρέπει να υπάρξουν πολύπλοκες λύσεις για την ανάπτυξη της Ευρώπης συνολικά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό τώρα έχει τον λόγο η κυρία Γκέντς. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Οι χώρες για τις οποίες μιλάμε είναι νέα κράτη-μέλη μετά την άλλαγη έπρεπε να φροντίσουν τα θύματα της άλλαγης ε, αυτής και να κάνουν διαρθρωτικές αλλαγές για να είναι ανταγωνιστικές σε μια ελεύθερη αγορά και να δημιουργήσουν νέες οικονομικές δομές. Και εδώ πέρα ε, οι πολίτες δεν έχουν και αποταμιεύσεις, δεν μπορούν να αποπληρώσουν τα στεγαστικά τους δάνεια και υπάρχουν όλο και περισσότερες δυσκολίες και όλο και περισσότερες κοινωνικές δαπάνες από πλευράς κυβερνήσεων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα αστάθεια η οποία εξαπλώνεται και μαζί με αυτήν εξαπλώνεται και ο λαϊκισμός. Όλα αυτά πρέπει να τα έχουμε κατά νου και να κινηθούμε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αλληλεγγύης. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριε κύριος Κλούτε τώρα έχει τον Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα το οποίο συζητάμε απόψε έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ως γνωστόν η Ευρωπαϊκή Ένωση προσανατολίζεται σε αυτά τα οποία λέει το, Ευρωπα... το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να δώσει εγγύησεις. Γι' αυτό ξανά και ξανά απευθύνει εκκλήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προς την Κομισιόν. Το Νοέμβριο του 2008 ζητήσαμε να αναλύσει τα αποτελέσματα της συμπεριφοράς των τραπεζών όταν ε, τους δώσαμε εγγυήσεις. Τον Απρίλιο, 24 Απριλίου φέτος επαναλάβαμε την ίδια έκκληση και μετά ζητήσαμε μία ανακοίνωση προθέσεων της Κομισιόν για το τι θα γίνει λεπτομερός όσον αφορά τις ενισχύσεις ε, αυτές και από όσο γνωρίζω δεν είχαμε καμία απάντηση μέχρι σήμερα. Οπότε το ερώτημα είναι πράγματι δεν έλαβαμε καμία απάντηση και αν ισχύει αυτό γιατί. Και το τρίτο ερώτημα πότε να περιμένουμε απάντηση σε αυτά τα ερωτήματά μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κλούτε για δύο λεπτά ο κύριος Στολόγιαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ κατάγομαι από μια χώρα η οποία έλαβε ενισχύσεις ε, δημοσιονομικές από την Κομισιόν, από τη Ρουμανία. Γι' αυτό θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για το ότι κινήθηκε τόσο γρήγορα για να δώσει αυτή την στήριξη στην Ρουμανία. Χωρίς αυτή την οικονομική στήριξη τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα θα είχαν οξυνθεί ακόμη περισσότερο. Βεβαίω υπάρχουν ε, πολλά κοινωνικά προβλήματα στις χώρες ε, που έλαβαν αυτή τη χρηματοδότηση και μπορούμε να συζητήσουμε το τι σημαίνουν αυτοί οι κοινωνικοί όροι που θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις ε, συμφωνίες αυτές. Εάν το δούμε όμως έτσι, πρέπει να λάβουμε υπόψη πως ε, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που υπάρχουν σε αυτές τις χώρες οδήγησαν σε ανισορροπίες ε, και γι' αυτό ακριβώς χρειάστηκε αυτή η οικονομική ενίσχυση. Οπότε αν να μιλάμε για κοινωνικές προϋποθέσεις πρέπει να μιλήσουμε οπωσδήποτε και για μεταρρυθμίσεις στον κοινωνικό τομέα πρώτα απ' όλα του τομέα των συντάξεων για να υπάρχει κοινωνική βιωσιμότητα μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπίσουμε τη ρίζα του προβλήματος. Ευχαριστώ. Για ένα λεπτό, κύριος Ντερόσα. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, Επίτροπε Αλμούνια, η ILO, η διεθνής, ε, το Διεθνές Γραφείο ε, Απασχόλησης Εργασίας, είπε ότι ε, η Ευρώπη θα μεταμορφωθεί προς το καλύτερο μετά την κρίση. Δυστυχώς δεν θα γίνει αυτό. Θα έπρεπε να έχουμε με πιο αηφόρα οικονομία, μια δίκαιη παγκοσμιοποίηση και μια εφαρμογή των στόχων της ναι. χιλιετίας. Δυστυχώς δεν οδεύουμε προς τα εκεί. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, οι χρηματοπιστωτικές δυνάμεις χαρακώνονται για να τηρήσουν τα προνομιά τους ενώ συγχρόνως αντλούνται εκατομμύρια, δισεκατομμύρια για την διάσωση τραπεζών. Τράπεζες όμως που καταστρέφουν τις ντόπιε πρωτοβουλίες και εμείς τις υποστηρίζουμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τις υποστηρίζει. Η υπηρεσία του Δουβλίνου δημοσίευσε σήμερα ένα έγγραφο μεταρρύθμιση στην ύφεση. Παραθέτω. Ιδανικά θα έπρεπε μέτρα για την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών να συνδυαστούν με μακροπρόθεσμους στόχους. Θα πρέπει η Κομισιόν να επιμείνει, αν μη τι άλλο, να προσπαθήσουν να το κάνουν αυτό τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ντερόσα. Περνάμε τώρα στο κύριο της οφθαλμοθυρίας. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Σεκέρσκι. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από την οικονομική κρίση, από βαριά οικονομική κρίση, τα κράτη-μέλη δικαιολογημένα ζητούν κάποια χρηματική βοήθεια. Το θέμα που τίθεται είναι ποιο τμήμα της βοήθειας αυτής φτάνει μέχρι τα χέρια όσων την χρειάζονται περισσότερο, δηλαδή των πιο ευάλωτων πολιτών. Θέσεις εργασίας γάνονται κάθε μέρα και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών λαμβάνουν άραγε υπόψη τους την κοινωνική πτυχή του προβλήματος όταν χορηγούν τη βοήθεια αυτή, όταν την κατανέμουν. Φροντίζουν να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας ή να ανυψώσουν το βιωτικό επίπεδο. Σας ρωτώ λοιπόν, σας ζητώ να μην κλείσετε τα μάτια στις ανάγκες των πιο ευαλώτων. Για ένα λεπτό τώρα... Για ένα λεπτό η Ευχαριστώ. Η εφαρμογή της αρχής της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής είναι ιδιαίτερα σημαντική σε καταστάσεις κρίσεως. Σημαντική αύξηση του κοινοτικού προπολογισμού μεν και ισότιμη κατανομή του κοινοτικού πλούτου δε κοινωνική συμπερίληψη, δημιουργία θέσεων απασχόλησης με δικαιώματα για όλους, πρόσβαση στις δημόσιες οικουμενικέ ποιοτικέ υπηρεσίες για να διασφαλιστούν τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών. Έτσι, όχι μόνο τα κοινοτικά χρήματα, αλλά και όλες οι προτάσεις για οικονομικές και χρηματοπιστωτικές ε, παρεμβάσεις θα πρέπει να αξιολογούνται από τις κοινωνικές συνέπειες που έχουν, τόσο ώστε να μην επιδεινωθεί η κατάσταση της ανισότητας και της ενδείας. Ας ελπίσουμε κύριε Επίτροπε ότι μετά από αυτή τη συζήτηση θα αναλάβετε πρωτοβουλίες προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κέλλη. Äh, Uh, ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε λέγω. Και ε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η απόψινή συζήτηση για τη δρακαλή πίστη η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει αυτές τις χώρες ε, που βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και το ζήτημα είναι το εξής όταν ε, διατίθεται τέτοια κονδύλια με αυστηρές ε, συνθήκες τι πρέπει να γίνεται πρέπει να διασφαλίσουμε πως ε, δεν θα έχουμε κάκο διαχείριση αυτών των χρημάτων Νομίζω, το είπε και η κυρία Χάρκιν, πως πρέπει να υπάρχει εμπιστοσύνη αμοιβαία και δεύτερον δεν θα φτάσουμε ποτέ στην κατάσταση που περιγράφει ο κύριος Ντερόζα του να έχουμε μια καλύτερη κατάσταση μετά την κρίση από ό,τι έχουμε τώρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέλλη. Ο κύριος Επιτρόπος. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ πλήρω στι προποθέσει και τα κριτήρια που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό κάνει και η Κομισιόν όταν δανείζει χρήματα σε αυτά τα τρία κράτη-μέλη με τη διευκόλυνση ισουσγείου πληρωμών. Αυτό κάνει. Δανείζει χρήματα υπό ακριβώ τι ίδιε προποθέσει και συνθήκε. Ευνοϊκότερε μεν από αυτέ που ισχύουν στην αγορά αλλά με προϋποθέσεις για την αποπλήρωση, για την εξυπηρέτηση του δανείου. Πάντως, το θέμα είναι ότι όταν χρησιμοποιείται αυτή η διευκόλυνση, το ισοζυγείο πληρωμών δηλαδή, του ισοζυγείου πληρωμών, η ενίσχυση, θα πρέπει να κάνουμε τη διάκριση μεταξύ μιας εξουσιοδότησης χρήσης κάποιων πόρων, διαθροτικά ταμεία, μία πέθρου κτλ. με τα μέτρα επίλυσης ενός οικονομικού ή χρηματοπιστωτικού ή δημοσιονομικού προβλήματος. Η Ρουμανία, η Λετωνία αναγκάστηκαν να στραφούν σε μας γιατί δεν μπορούσαν να στραφούν αλλού. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μιλάμε για χρήματα για ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, για μια συγκεκριμένη δραστηριότητα. Όχι. Μιλάμε για χώρες που έχουν δημοσιονομική δυσκολία που εν μέρει οφείλεται στην κρίση αλλά που είναι πολύ οξύτεροι από χώρες που πλήττονται από την ίδια κρίση λόγω κακοδιαχείρισης. Και παρακαλώ μην θεωρήσετε που δεν είναι υπεύθυνη ούτε την Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο των Υπουργών για την κακοδιαχείριση ορισμένων κυβερνήσεων ορισμένων κρατών μελών. Δεν είναι δική μας ευθύνη. Αυτή η ευθύνη μας είναι να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε να επιληθεί ένα δημοσιονομικό πρόβλημα. Δημοσιονομικό πρόβλημα σημαίνει εν μέρη πρόβλημα ισοζυγίου πληρωμών. Χρέους. και εν μέρη είναι ανάγκες του δημοσίου. Σε αυτή την περίπτωση, για το δημόσιο χρέος δηλαδή, έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε κάποιες συγκεκριμένες προϋποθέσεις και όρους. Αυτό κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Προχθές, την τρίτη, την τρίτη εδώ στις Βρυξέλλες, ακόμα προσπαθούσα να πείσω έναν εκπρόσωπο της λετωνικής κυβέρνησης τα μέτρα που θα συμπεριλάβουν στον προπολογισμό του του 2010 να είναι πιο προοδευτικά. Μην ζητάτε όμω από την Κομισιόν να υποχρεώσει μια χώρα να εφαρμόσει ή να εγκρίνει μια ε, φορολογική μεταρρύθμιση που δεν θέλει να εγκρίνει, που δεν θέλει να περάσει. Τι εναλλακτική έχουμε στο όνομα των ε, Ευρωπαίων πολιτών. Να αφήσουμε αυτές τις χώρες να φαλυρίσουν να υποτιμήσουν κατά 25 ή 30% το εθνικό τους νόμισμα. Κάτι το οποίο σήμαινε ότι θα είχε λιγότερα λεφτά στην τσέπη του ο απλός πολίτης. Εγώ συμφωνώ με την αναλύση σας. Αυτά που είπε ο κ. Ντερόσα, ο κ. Στέρκας, όλοι σας. Συμφωνώ, κλά, ε, σαφώς. Αλλά χώρες όπως η Ρουμανία, όπως ε, η Λετωνία αντιμετωπίζουν πιο πολύπλοκη πραγματικότητα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, δεν είναι μανιχαϊστικά όλα, άσπρα ή μαύρα. Μπείτε στη θέση μας, στο κάτω-κάτω. Δεν μπορούν να δανειστούν από τις αγορές αυτές οι χώρες. Σε ποιον θα στραφούν, αν δεν μπορούν να στραφούν σε εμά. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι έχουν τα πράγματα. Και αυτό προσπαθούμε να κάνουμε υπό τις ε, προϋποθέσεις με τις οποίες βεβαίως και εσείς συμφωνείτε. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ. Κύριε Αλμονία, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε αυτό το σημείο και πάμε στη δήλωση της Επιτροπής για την πολιτική κατάσταση στην Ομδούρα εν ώψη των εκλογών στη χώρα. Το λόγο έχει. Ας αφήσουμε τους επιτρόπους να φιλήσουν.